Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση αρχικά. Η οποία έχει ως εξής. Σύμφωνα με το άρθρο 166 του κανονισμού, ο πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει ποινή στον κύριο Ντεκράφ για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της 28 Οκτωβρίου 2015 αυτό αφορά πενθήμερη αποζημίωση και ε, είναι γνώση ε, του κυρίου Τεγράφη η απόφαση αυτή για πενθήμερη ε, παρακράτηση αποζημίωσης. Λοιπόν, θα μιλήσω ρουμανικά.